Bardzo proszę. Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το τμήμα της συνεδριάσεως που αφορά κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Να σας πω ότι έχουμε ήδη δύο ώρες εδώ, αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Έγκριση ημερησία διατάξεως φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό. Ε, να σας πω ότι έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες και ότι μεταδίδεται μέσω διαδικτύου η συνεδρίασή μας. Τώρα θα συζητήσουμε σχετικά με την ανταλλαγή απόψεων για την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις νέες τεχνικές ε, αναπαραγωγής. Θα, κάνουν, θα γίνει μια μικρή ε, εισαγωγή και μετά θα δώσω τον λόγο στον κύριο Νίλ Στόρβαλα ε, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα μιλήσουμε λοιπόν ε, για την απόφαση του δικαστηρίου για τις νέες τεχνικές αναπαραγωγής. New Breeding Techniques. Πρόκειται για ένα αίτημα το οποίο έχει υποβληθεί από την Επιτροπή μας και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος επίσης καθότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αφορά και τις δύο ε, επιτροπές μας και ενδιαφέρει και τις δύο επιτροπές εξίσου. Εξού λοιπόν και αυτή η κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου ΕΦΕΝΟΣ και Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας Ασφάλειας Τροφίμων αφετέρου. Ε, στις 25 Ιουλίου του 2018 το δικαστήριο απεφάνθη ότι οι οργανισμοί οι οποίοι προκύπτουν από την μεταλλαξογένεση είναι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί και επομένως διέπονται από τα όσα αναφέρονται στην οδηγία ε, για τα, ε, τους μεταλλαγμένους οργανισμούς. Ορισμένοι διατείνονται ότι οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να περνούν από διαδικασία αδειοδότησης που και μακρά είναι και ε, κοστίζει. Ενώ υπάρχουν άλλοι που λένε ότι θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επενδύσουν στον τομέα αυτό. Οπωσδήποτε θα πρέπει ε, να ε, υπάρξουν διευκρινιστικές αρχές έτσι ώστε και επεξηγήσεις έτσι ώστε οι εμπλεκόμενοι στον τομέα αυτό να ξέρουν που βαδίζουν. Κύριε Τερβάλε, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Γεωργίας και σας δίνω μέσω το λόγο. Συμπτώσεις πολλές συμβαίνουν στη ζωή. Την ημέρα των ε, Αθών αποφάσισα ε, να πάω στην Στοκχόλμη και να περάσω τα Χριστούγεννα με τη γυναίκα μου που δεν με έχει δει και πολύ τον τελευταίο καιρό. Και το πρώτο που έκανα όταν έφτασα στην ε, Στοχόμη, ε, άνοιξα την τοπική εφημερίδα και ε, είδα ένα άρθρο ενός καθηγητού από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Το ενδιαφέρον λοιπόν με το άρθρο αυτό ήταν ότι αμφισβητούσε τη σοφία ε, του ε, δικαστηρίου. Και γιατί, διότι το σημείο εκκίνησης ήταν ότι το 2050 θα έχουμε δύο δις ε, κατοίκους στον κόσμο. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να τραφούν με κάποιο τρόπο. Και εάν δεν έχουμε μια ικανή γεωργία, δεν θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε όλους αυτούς ε, τους ε, ε, ανθρώπους. Από εκεί ξεκινούσε λοιπόν και μετά προχωρούσε σε μία συζήτηση σχετικά με την τεχνολογία DNA. Ε, αυτά, αυτή την θεωρία για τα ψαλίδια, το ψαλίδισμα του DNA μέσω του οποίου μπορείς να δημιουργήσεις κάτι καινούριο. Η απόφαση του δικαστηρίου άφησε όμως ανοιχτό το ζήτημα αυτό. Και έβαλε και τη Γεωργία ε, σε δύσκολη θέση. Γιατί είναι δύσκολο να έχεις ανταγωνιστική γεωργία με τέτοιες συνθήκες, στην Ευρώπη πάντα. Αναφέρθηκε λοιπόν και σε κάτι άλλο, ότι έχουμε την τάση να μοιραζόμαστε ε, την ε, πληροφόρηση με διαφορετικό τρόπο. Και διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στην πραγματική ζωή οι ακτιβιστές, ε, τα άτομα γενικά, ακολουθούν ε, και ενστερνίζονται κάποια στοιχεία της ε, επιστημονικής προσέγγισης, αλλά αφήνουν ε, απ' έξω κάποια άλλα στοιχεία της απονομιστικής επιστημονικής προσέγγισης. έξω και η παράνοια που προκύπτει και, επομένως, γι' αυτό ακριβώς προκύπτει και η ανάγκη εντελεχούς εξετάσεως της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικοστηρίου, έτσι ώστε να ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, όχι μόνο για μας τους Ευρωπαίους, αλλά και για όλους τους κατοίκους του πλανήτη που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τραφούν. Δεν είμαστε μόνο εμείς η Ευρώπη, αλλά εάν δεν είμαστε εμείς αρκετά ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο, τότε δεν θα καταφέρουμε ούτε να ε, θρέψουμε τους εαυτούς μας, άρα θα δημιουργηθούν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Άκουσα κάποια σχόλια από την πλευρά των πρασίνων ε, και αυτό με προειδεάζει για μια πάρα πολύ ζωντανή συζήτηση. Ε, Βεβαίω το θέμα δεν θα ολοκληρωθεί και η συζήτηση επί του θέματος δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα, αλλά μερικές φορές λέω ότι πρέπει να δεχτούμε την πραγματικότητα έτσι όπως έρχεται. Ευχαριστώ. Ωραία λέει ο Πρόεδρος. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις εγωγικές παρατηρήσεις. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο σε έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, πρόκειται για την κυρία Σαμπίν Γιούλιχερ. η οποία θα μας μιλήσει για αυτή την απόφαση του δικαστηρίου και μετά θα δώσουμε το λόγο εις τους βουλευτές. Ε, ε, παρακαλώ πολύ την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ και καλό απόγευμα σε όλους. Καλή χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω τις δύο επιτροπές που οργάνωσαν αυτή την ανταλλαγή απόψεων για το αποτέλεσμα της απόφασης του δικαστήριου. Είναι ενδιαφέρον για μας, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ακουστούν οι απόψεις σας. Λοιπόν, τι έκανε το δικαστήριο. Το δικαστήριο διευκρίνησε το πεδίο της νομοθεσίας περί γάμματα για κάποιες τεχνικές. Σε ό,τι αφορά τις, α, τεχνικές αυτές, τις, μεταλλαξιογόνες. Δεν αλλάζει κάτι όμως στον ίδιο τον κανονισμό. Το δικαστήριο διευκρίνησε ότι η νέα νομοθεσία γραμματοφωνικών αφορά προϊόντα τα οποία προέκυψαν και από νέες τεχνικές μεταλλαξιογόνες και θα πρέπει οι επιχειρήσεις να, εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τα οποία διατίθεται στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός είναι ασφαλή και αφετέρου συμμορφώνονται με τις απαιτήσει. Και τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για να ελέγξουν και να υλοποιήσουν αυτές τις διατάξεις. Μετά από την απόφαση αυτή του Ιουλίου, πέρσι η Κομισιόν οργάνωσε μια σειρά από ε, επαφές με τις ε, Εθνικές Αρμόδιες Αρχές στα πλαίσια της Μόνιμης Επιτροπής που είναι υπεύθυνη για αυτήν την νομοθεσία και συζητήσαμε με τα κράτη-μέλη και θυμήσαμε στα κράτη-μέλη την ευθύνη που έχουν να εφαρμόσουν την νομοθεσία περί γάμματα φόμικραν σύμφωνα και με την απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, μιας και τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο. Αυτό περιλαμβάνει και τη συμμόρφωση με την νομοθεσία γάμματα φόμικρων, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά στην, της Ευρωπαϊκής και σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με βάση τις δοκιμές που λαμβάνουν χώρα τις ε, τωρινές και τις μελλοντικές. Είναι δύο οι πτυχές. Ε, στις συζητήσεις αυτές, στις συναντήσεις με τους εμπειρογνώμονε των κρατών μελών, μοιραστήκαμε κάποιες πληροφορίες, ε, υπόθηκε ότι υπάρχουν κάποιες προκλήσεις στην εφαρμογή αυτής της απόφασης του δικαστηρίου, για να είμαι σαφής, ε, το πρόβλημα δεν είναι τόσο να καταλάβουμε την απόφαση, αλλά το πώς θα την εφαρμόσουμε. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις όσο χρειαστεί, ε, για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εφαρμόσουν αυτήν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ίσως είναι και η μεγαλύτερη ε, σε επίπεδο εφαρμογής, και θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα αυτό εδώ μετά για τη συζήτησή μας, ε, υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία είναι παρόμοια, τα οποία όμως έχουν προκύψει από διαφορετικές τεχνικές επεξεργασίες και ανάλογα με την τεχνική με την οποία φτάσαμε στο προϊόν αυτό, μπορεί αυτά τα προϊόντα να εμπίπτουν σε διαφορετικά αριθμιστικά καθεστώτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ε, για να ελέγξουμε και να εφαρμόσουμε την νομοθεσία πρέπει να μπορούμε να διαφοροποιήσουμε, να ξεχωρίσουμε τα προϊόντα που ε, βασίζονται σε μια συγκεκριμένη τεχνική, έχουν παραχθεί βάσει μια συγκεκριμένη τεχνική. Αυτή είναι μια πρόκληση. Ε, έτσι λοιπόν η Κομισιόν ζήτησε από τα το, ευρωπαϊκά εργαστήρια αναφοράς για τους γραμματοφόμικρων να εξετάσουν αναλυτικά τις προκλήσεις αυτές και τις ενδεχόμενες λύσεις. Αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης τον Μάρτιο Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω ότι αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται να λάβει η χώρα κάποια αξιολόγηση της νομοθεσίας φόμικρον. Ούτε να υποβληθεί κάποια νέα νομοθετική πρόταση τουλάχιστον κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως θα πρέπει μέσω μακροπρόθεσμα και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα σύστημα διακυβέρνηση που ε, θα παρακολουθεί τι εξελίξει, δεν θα μένει πίσω, σε επιστημονικό επίπεδο ενώ, και ταυτόχρονα ε, θα ε, ε, προωθεί την υπεύθυνη καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και θα εξασφαλίζει και την ασφάλεια. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις σε κοινωνικό επίπεδο, κάποιες αναφέρθηκαν ήδη, υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει ανάγκη ενός βιώσιμου συστήματος γεωργοδιατροφικού. Το θέμα είναι κατά πόσο το ρυθμιστικό πλαίσιο του ΓΑΜΑΤΑΦΟΜΕΤΡΟ και το σύστημά μας είναι αρκετά ανθεκτικό για να αντιμετωπίσει αυτές τις αλλαγές που προκύπτουν, τις επιστημονικές, τις νέες τεχνολογίες και ταυτόχρονα να επιτεχάνεται ο στόχος σχετικά με την ασφάλεια και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Όπως γνωρίζουμε από το παρελθόν, από τις πολλές συζητήσεις που είχαμε και εδώ και αλλού, ξέρουμε ότι είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι δημιουργεί αντιπαράθεση. Κατά την άποψή μα, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει ένα ανοιχτό, ειλικρινή διάλογο με όλου του εμπλεκόμενου η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει μια σαφή εικόνα αφενός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και από τα κράτη-μέλη για το τι θεωρείται ότι πρέπει να είναι το μέλλον ε, της ευρωπαϊκής βιοτεχνολογίας και τι αλλαγές πρέπει να λάβουν χώρα μέσω μακροπρόθεσμα. Αυτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τη δυνατότητα που μας δώσατε να κάνω αυτή τη δήλωση και αναμένω να ακούσω και την ανταλλαγή απόψεων που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, ένα αίτημα παρακαλώ λέει ο Πρόεδρος. Πρέπει να ζητήσετε το λόγο γρήγορα για να ξέρουμε πόσοι θέλουν το λόγο και να μοιράσουμε και τον χρόνο μιλίας πιο αποτελεσματικά. Ξεκινάμε με τον κύριο Άγνιου. Νομίζω ότι θα έχουμε 1,5 λεπτό καθένας. Κύριε Άγνιου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 115 περίπου ευρωβουλευτές συμμετέχουν στην Άγκρη και στην Ένβη. Μπορεί να είναι και 100 εδώ. Θα μπορούσαν να είναι 100 εδώ, αλλά είναι 20. Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Ε, πραγματικά θα μπορούσατε να καταλάβετε καλύτερα αν σας μιλούσα για τα τρακτέρ. Τα τρακτέρ ε, πήραν τη θέση των ε, αλόγων, έσπροχναν απλώ. Μετά δημιουργήθηκαν νέες τεχνολογίες. Ε, το ίδιο ε, έλεγαν τότε κάποιοι ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τέτοιες νέες τεχνολογίες. Ε, ε τι θα έχει γίνει τότε. Θα πρέπει να εισαγάγουμε τώρα τρακτέρ. σε αυτή την νομοθεσία ε, πραγματικά στην Αγγλία δεν μπορούμε να πιστέψουμε πώς έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί. Άλλο γενετικό τροποποιημένο, ε, άλλο γενετική επεξεργασία. Ε, στη γενετική επεξεργασία απλά ε, δίνουμε μια όθηση σε μια μετάλλαξη η οποία όμως γίνεται φυσικά, δεν, δεν προσθέτουμε DNA από αλλού. Εγώ συμμετέχω στη Γεωργία από το 1971. Ε, έχω δει τις διάφορες τεχνικές, ε, το ζευγάρωμα, το τυχαίο, ε, αυτό δεν μας πάει πολύ μακριά. Μετά έχουμε την επιλεκτική εκτροφή στο ίδιο είδος, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση και μετά είδαμε ότι μπορεί να υπάρξει μετάλλαξη φυσική, αυτό μας έδωσε μια ευκαιρία. Αυτό που προσπαθούν να κάνουμε, να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, είναι να, αυτή την ευκαιρία να την εκμεταλλευτούν, να την διαχειριστούν, να την ελέγξουν. Εάν αυτό προχωρήσει, ναι, αυτό είναι, αυτό, το, αυτή η νομοθεσία προχωρήσει, τότε τέρμα αυτή η προσπάθεια και θα τα, θα τα αναγκαστούμε να τα εισάγουμε όλα αυτά στο μέλλον. Δεν έχει κανένα νόημα, είναι χαζό και πρέπει να, να αναστραφεί αυτή η νομοθεσία. Ο κύριος Αντρίο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε να πω και εγώ δύο λόγια. Ε, θεωρώ ότι το δικαστήριο στην απόφαση αυτή επιδεικνύει μεγάλη σοφία έτσι το ελαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον διότι μας λέει ότι οι τεχνικές αυτές μετάλλαξεις περιλαμβάνουν κάποιους κινδύνους, κάποιο ρίσκο. Όπως είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, το, με, το μέλλον των βιοτεχνολογιών πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μια μεγάλη συζήτηση και θα ήθελα στην επόμενη θητεία να έχουμε τη δυνατότητα να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Διότι το διακύβευμα είναι μεγάλο. Από τη στιγμή που υπάρχει κίνδυνο όμω, που υπάρχει ρίσκο, η εμπειρία μα δείχνει ότι πρέπει ε, ανάμεσα στα συμφέροντα των μεγάλων βιομηχανιών, το περιβάλλον, τη διατροφή, ε, δεν είναι πάντα ίδιοι στόχοι ε, ανάλογα με το που, από πού το βλέπει κανεί. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα ζητήματα βιοπικιλότητα, τα ζητήματα του κλίματο, τα ζητήματα τη υγεία που πρέπει να είναι στην καρδιά των συζητήσεών μα, πρέπει να μα οδηγήσουν να σκεφτούμε την ευθύνη που έχουμε στον τομέα τη βιοτεχνολογία. Που όπω και να έχουν τα πράγματα, θεωρώ ότι η, απόφαση του δικαστηρίου είναι εξαιρετικά υπεύθυνη, είναι σοφή και είναι στο ύψο των ε, του διακυβεύματος θα έλεγα. Ευχαριστώ. Κύριε Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει, αλλά είναι λίγο περίεργο το γεγονό ότι γίνεται με τοπική επίθεση από τα έδρανα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Την απόφαση αυτή θα πρέπει να την ε, δεχτούμε. Είναι απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό μπορεί να μην μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, αλλά το να λέμε ότι θα πρέπει να αλλάξει ο νόμο, αυτό θεωρώ ότι είναι με τοπική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τι αποφάσισε το δικαστήριο. Σαφή επισήμανση να ελέγχονται όλα αυτά ενδελεχώ και να εκτιμάται ο κίνδυνο τη τεχνολογία. Νομίζω ότι και τα τρία αυτά στοιχεία έχουν να κάνουν κάτι με την προστασία της του ε, καταναλωτή και την αρχή της πρόληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιο ε, με το επιθυμεί αυτή, τουλάχιστον θα πρέπει να αποδεχτεί την προστασία του καταναλωτή. Αλλά γι' αυτό είναι πολύ σωστή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σοφή γιατί είναι προς το συμφέρον του Ευρωπαίου καταναλωτή. Στο επίκεντρο λοιπόν είναι η σωστή επισήμανση για να ξέρει ο καταναλωτής τι τρώει στο πιάτο του. Το να λέμε τώρα ότι θα πεθάνουμε όλοι από την πείνα είναι θεωρώ απόλυτη ανοησία. Ανοησία. Να κοιτάξουμε τι έγινε και πριν από 20 χρόνια όταν έγινε η συζήτηση με την προηγούμενη γενετική τεχνολογία. Βλάφτηκε τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις τεχνολογίες αυτές. Δεν ήταν κάποια τέτοια αποδυνάμωση των αγορών. Αντιφετέω, οι ΕΠΑ εισαγάγουν ευρωπαϊκά τρόφιμα γιατί δεν έχουν αρκετά δικά τους. Γι' αυτό λοιπόν όλες αυτές οι προβλέψεις της Κασάνδρας για την ευρωπαϊκό σκηνικό είναι θεωρώ ανοησία. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν θέλουν γενετική τεχνολογία αυτό το έχουν πει και στους παραγωγούς και στους αγρότες. Και σε αυτό θα πρέπει να προσαρμοστούν οι αγρότες και οι παραγωγοί. Και γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζω την απόφαση αυτή του δικαστηρίου. Μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να συνταχθούμε με την απόφαση αυτή και θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη σήμανση και στις εισαγωγές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βάιτς, λέει ο πρόεδρος. Δεν θα είμαι τόσο μετριοπαθής όπως ο συνάδελφος έρχεται ένας ε, ε, εκπρόσωπος της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος για να μας απευθύνει τέτοιες ρητορίες της, της βιομηχανίας. Αυτό είναι απόλυτη ανοησία. Η Ευρώπη καλύτερα να θέλει τον κόσμο και ξέρουμε ότι υπάρχει διάβρωση Υπάρχει αλάτωση του εδάφου. Χρειαζόμαστε λοιπόν βιώσιμα μοντέλα καλλιέργεια, όχι ακόμα πιο πολύ γεωργική βιομηχανία. Δεν ξέρω πώς βγαίνετε και τα λέτε αυτά που λέτε. Πέραν αυτών, πιστεύω ότι οι επιπτώσει ε, των δίθεν ε, επακριβόλων αυτών τεχνολογιών είναι πολύ αμφιλεγόμενες. Υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις ότι υπάρχουν πολλές ανεπιθύμητες παρενέργειες οι οποίες θα τις πληρώσουν τελικά οι επόμενες γενιές και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τους γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί να παράγονται στη φύση, όχι στα εργαστήρια. Αυτή η επιχειρηματολογία που προβάλλεται είναι πραγματικά ε, περίεργη. Και τι να σας πω, αυτή είναι η δημοκρατία. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θέλουν να ξέρουν τι αγοράζουν και τι τρώνε. Αυτό λοιπόν πρέπει να ικανοποιήσουμε ω έτοιμα και προς την κατεύθυνση αυτή οδεύει η δικαστική αυτή απόφαση και το αν το αμφισβητείτε αυτό θεωρώ ότι αμφισβητείτε την ίδια την δομή της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ περίεργο. Ο πρόεδρο. η Δημοκρατία είναι η δυνατότητα να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις οι οποίες να υφίστανται. Ο κύριος Χάδημα, ευχαριστώ. Ε, πολύ, Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ συναισθηματική και πολύ δογματική τελικά εκτελήσεται και όχι αντικειμενική όπως θα έπρεπε. Είναι κρίμα αυτό. Να το κοιτάξουμε με πιο αντικειμενικό τρόπο. Εγώ πιστεύω πάντα ότι για να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά και για να βελτιώσουμε τη βιωσιμότητα της γεωργίας μας η εκτροφή και η είναι απαραίτητη και δεν μπορούμε να την ε, αμελήσουμε. Ε, και θα πρέπει λοιπόν με αυτή την τεχνητή τροφή να, να επιλύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ο τομέας της γεωργίας αυτής, της βιολογικής ε, γεωργίας προσπαθεί να αντιμετωπίσει προβλήματα. Αυτός ο πολλαπλασιασμός λοιπόν χρησιμοποιείται με νέους ε, τρόπους. Διαφωνώ μαζί σας ε, ότι η νομοθεσία είναι περίεργη και αντιφατική. Γιατί αυτό που επιτρέπεται, επιτρέπεται και συμβατικά. Βάζουμε μια ατομική, λοιπόν, ατομική βόμβα σε μια, σαν ένα και δημιουργείται μια μετάλλαξη, την οποία και χρησιμοποιούμε με κάποιον τρόπο και τελικά αυτό μας οδηγεί σε πλανεκτήματα. Δεν επιτρέπεται όμως στοχευμένη τέτοια μετάλλαξη από την ομόθεση. Αυτό είναι περίεργο. Από το 2001 και μετά το παράρτημα των νέων τεχνικών γειτονικής αναπαραγωγής δεν έχει προσαρμοστεί. Όλοι ξέρουμε ότι έχει αλλάξει ο κόσμος, όλοι ξέρουμε ότι οδεύει ταχαίως και προχωράει ταχαίως η επιστήμη, η γνώση. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να γίνει μια διαφορετική συζήτηση, να το κοιτάξουμε το θέμα λίγο πιο αντικειμενικό και πραγματικό τρόπο, πραγματιστικό τρόπο. Τι τεχνικές αναπαραγωγής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με δεντολογικό τρόπο, να τις δεχτούμε ηθικά, αν θέλετε, και να δούμε και τα τα πλεονεκτήματα για τη βιωσιμότητα, για την ε, ενοποιημένη διαχείριση αποβλήτων. Να κοιτάξουμε λοιπόν το 2001 τι έγινε. Και τέλος, αν δεν κάνουμε τίποτα και μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα τελικά, μόνο οι πολυεθνικές, οι μεγάλες πολυεθνικές θα χρησιμοποιούν αυτές τις ε, ε τεχνικές αναπαραγωγής ε, και του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού, γιατί αυτέ μπορούν να ελέγξουν την νομοθεσία και οι μικρέ τελικά επιχειρήσει, οι οποίε και έχουν να τα χρησιμοποιήσουν όλα αυτά, δεν θα μπορούν να το, να το κάνουν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι ε, οι οργανισμοί οι οποίοι προέρχονται από μεταλλαξογέννηση εμπίπτουν εις το, στην οδηγία ε, για τους γάμματα φόμικρον. Όμως αυτή η διαδικασία ε, παραμένει η μόνη δυνατότητα που έχουν όσοι πολίτες αρνούνται ε, τα, την καλλιέργεια μεταλλαγμένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες δέχονται ε, τα μεταλλαγμένα και προωθούν και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Επομένως, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν τα μεταλλαγμένα, παρόλα αυτά ε, ε, πρέπει να τα υποστούν κυρίως λόγω ε, των εμπορικών πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεταλλαξογένεση μπορεί να είναι φυσική ή όχι, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, δεν είμαι και ειδικό άλλωστε, αλλά η φυσική μεταλλαξογένεση δεν εμπίπτει στο θέμα των γάμα τάφα άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ξεκαθαρίσουμε για ποιο είδος μεταλλαξογέννησης μιλάμε ε, εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να πούμε ότι ε, δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε μια τέτοια κατάσταση. Εμείς ε, θεωρούμε ότι η απόφαση είναι σωστή και είναι δικαιολογημένο και το νομικό πλαίσιο, έστω και αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση του και τον νόμο του 2014 στη Γαλλία. Επομένως, θεωρούμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, δεχτούμε αυτές, ε, αυτούς τους περιορισμούς, έστω και αν καταλαβαίνουμε την αντίδραση κάποιων παραγωγών, παραγωγών που θεωρούν υπερβολικές, ε, υπερβολικούς αυτούς τους περιορισμούς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μακιντάιερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρώπη ήταν πρωτοπόρα στις αναπαραγωγικές τεχνικές. 50% της έρευνας ε, για αυτές τις τεχνικές ε, γίνεται στην Ευρώπη και μας είναι ιδιαίτερος ε, προσφυλής ε, και επομένως δεν είναι δυνατόν να πετάξουμε αυτό, αυτή την εμπειρία. Ε, στον σημερινό κόσμο έχουμε πολλές προκλήσεις. Την σπανιότητα των πόρων, την κλιματική αλλαγή, την αύξηση του πληθυσμού και επομένως οι επιστημονικές εξελίξεις είναι αυτές οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν να παράγουμε φυτά ε, για την κατάλληλα για την νέα εποχή. Αυτή τη στιγμή ε, μέσω των ε, μεθόδων που γνωρίζουμε μπορεί να χρειαστούν 18 χρόνια για να αναπτυχθεί ένα νέο είδος χλώης. Θέλουμε υλικό το οποίο δεν θα χρειάζεται ε, πολύ φροντίδα, δεν θα χρειάζεται πολύ νερό, που θα είναι πιο ανθεκτικό, που δεν θα χρειάζεται πολλά ζανιοκτώνα. Στο Ρόθεμστεντ έχουμε ένα Ινστιτούτο που κατάφεραν να δημιουργήσουν ε, ε, φυτά τα οποία παράγουν ωμέγα 3 αντίστοιχα με τα ωμέγα 3 των ε, ηχθιελαίων και μάλιστα χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες από μια χωματερή. Η επιστημονική κατανόηση και γνώση, έτσι όπως αναπτύσσεται, είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν είναι δυνατόν οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι μικρές μεσαίες ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις ε, να μείνουν έξω από αυτές τις ε, δυνατότητες και να αποκοπούν από τις δυνατότητες αυτές. Βεβαίως οι κτηνοτρόφοι μας, οι γεωργοί μας μόνο φτωχότεροι θα γίνουν αν μείνουν έξω από αυτές τις διαδικασίες. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οπωσδήποτε το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και χρειαζόμαστε πολύ χρόνο για να, το αντιμετωπίσουμε. Άλλωστε δεν, ε, ε, δεν σχολιάζονται ή μη μόνον εφαρμόζονται οι αποφάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μπορούμε όμως να πούμε ότι ενδεχομένως θα προκύψουν κάποιες διαφορετικές ερμηνείες ανάμεσα στην ε, τεχνική της ε, ε, μεταλλαξογένεσης και της τρανσγένεσης. Πρόκειται για διαδικασίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Έχουμε 17 χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν εθνικούς κανόνες που απαγορεύουν την ε, ε, χρήση και καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Αλλά άλλο είναι να χρησιμοποιήσει κανείς την μεταλλαξογένεση που μεταφέρουν, μετατρέπουν γονίδια. Ε, δεν είναι ίδιο, λέω, με κάποια στοιχεία τα οποία απλώς εμπλουτίζουν το DNA των φυτών και δεν έχουν πρακτικές φραγκεστάιν που τροποποιούν ε, το DNA των φυτών. Η γενετική ε, έρευνα ε, θέλει να δημιουργήσει ποικιλίε όπως ας πούμε υπάρχουν στον, ε, ε, στον αμπελοϊνικό τομέα που βοηθούν στη δημιουργία ποικιλιών πιο ανθεκτικών. Αυτές οι ποικιλίε είναι ποικιλίε οι οποίες έχουν επιτευχθεί από το γενεολογικό υλικό ε, της, ε, ε, του φυτού. Δεν είναι λοιπόν καθόλου μεταλλαγμένο προϊόν. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Δεν είναι μεταλλαγμένος ο οργανισμός, η κυρία Γκουανέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οπωσδήποτε οφείλουμε να χαιρετήσουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ορίζει ως ε, μεταλλαγμένους τους οργανισμούς που έχουν προκύψει από μεταλλαξογένεση. Βεβαίως ο καθένας έχει, δικαίωμα, ε, να, ε, έχει το δικαίωμα να επιλέγει τα τρόφιμα τα οποία θα αποτελέσουν την διατροφή τους. Ωστόσο υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι ε, προσπαθούν ε, υποτίθεται για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις των καιρών, να χρησιμοποιήσουν την βιοτεχνολογία. Αλλά η βιοτεχνολογία δεν είναι η μοναδική απάντηση ε, στις νέες προκλήσεις. Έχουμε την βιώσιμη γεωργία, έχουμε την εναλλακτική γεωργία, πρακτικές οι οποίες εξίσου μπορούν να αποτελέσουν λύσεις στο πρόβλημα ή στις προκλήσεις. Το δικαστήριο καταδεικνύει ότι είναι δυνατόν να ε, ε, θεωρήσουμε ε, γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς που έχουν προκύψει από μεταλλαξογένεση και αυτό σε αντίθεση με τα όσα ε, ανέφερε η βιομηχανία. Ε, η μεταλλαξογένεση ε, εμπεριέχει κινδύνους ε, και αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές πριν από οποιαδήποτε διάχυση της τεχνολογίας αυτής. Οπωσδήποτε δε θα πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη σήμανση και η χνηλασιμότητα καθώς επίσης και εμπορική παρακολούθηση αυτών των οργανισμών. στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο για την έκθεση Ζόμερ είχαμε την ε, δυνατότητα να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά τους ελέγχους. Πιστεύω λοιπόν ότι και για τις μεθόδους αναπαραγωγής ε, θα πρέπει και τις αναπαραγωγικές τεχνικές θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος. Ευχαριστώ η κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ πολύ. Όπως και άλλοι συνάδελφοι είπαν ότι ε, είναι εδώ μια συζήτηση η οποία είναι περισσότερο δογματική και λιγότερο ρεαλιστική. Έχουμε δηλώσεις οι οποίες στην ουσία έχουν ε, πρόσημο δεοντολογικό ή ηθικό ε, και όχι πρόσημο επιστημονικής αξιολόγησης. Πιστεύω ότι και εδώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο συνάδελφος Δεκάστρο. Ε, δηλαδή ότι να πούμε ότι εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ δεν θέλω να, ε, ε, να ερμηνεύσω οποιαδήποτε ή να σχολιάσω οποιαδήποτε απόφαση η οποία πρέπει να εφαρμοστεί. Όμως πιστεύω το εξής. Εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. δεν είναι το ίδιο η μεταλλαξογένεση και η τρανς γένεση. Επομένως ε, θα εφαρμοστούν συνολικά ε, ε, και χωρίς διαχωρισμό όλες αυτές οι αρχές επειδή δεν υπάρχει η αντίστοιχη κατάλληλη νομοθεσία όμως οι διαδικασίες δεν είναι καθόλου ίδιες. Ε, ε ίσως χρειάζεται κάποια νομοθέτηση ε, έτσι ώστε να αποφευχθεί ή να σταματήσει αυτή η σύγχυση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε λιγότερο δογματικοί, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία και οπωσδήποτε να διατηρηθούν όλα τα εχέγγυα της ε, διατροφικής ασφάλειας. Εγώ ξέρω ότι οποτεδήποτε γίνεται αναφορά ε, σε γάμα ταφ μικρόν ε, είναι ε, σαν να είναι ο διάβολος αλλά στην ουσία ε, πίσω υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία marketing γιατί όταν βάζει κάποιος στη συσκευασία ότι πρόκειται για προϊόν χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς αυτό το προϊόν αμέσως προωθείται πιο εύκολα. Ευχαριστώ. Ναι, Ακούστε, ένα μεγάλο μέρος ε, αυτών των μεταλλαξογενειογόνων ε, προέρχεται από επικίνδυνες ε, πηγές λένε κάποιοι, αλλά το δικαστήριο Φέντρο δεν συμφωνεί. Λέει ότι αυτή η τεχνική δεν αποτελεί γαματαφόμικρον, υπόκειται όμως σχετικές υποχρεώσεις. Αυτή η νέα λοιπόν γενιά γενετική μηχανική, η οποία από την δημιουργία αντιπαράθεση πρέπει να ελέγχεται. Θα πρέπει να ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και να περιορίζεται. Οι τροποποιήσει, ε, δηλαδή οι μεταλλάξει ζώων, ζωικών κυτάρων ή φυτικών κυτάρων πρέπει να ελέγχεται. Ποιε είναι οι επιπτώσει για το περιβάλλον, ποιε είναι οι επιπτώσει για ανθρώπινη υγεία, όπω και ε, για τι γάμματα φόμικρο. Εγώ προέρχομαι από την Κροατία. Η Κροατία είναι μια χώρα όπου απαγορεύονται οι γάμματα φόμικρον προσωπικά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαγορεύσει συνολικά τους φόμικρων και πρέπει η παραγωγή μας να βασίζεται στην ποσότητα και όχι στην αυξανόμενη στην ποιότητα και όχι στην αυξανόμενη ποσότητα ε, διότι η προστασία της ποιότητας είναι αυτή που θα μας κάνει και πιο ανταγωνιστικούς σε σχέση με άλλες αγορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι σημαντική αυτή η συζήτηση, αλλά βεβαίω ο καθένα λέει τη γνώμη του. Ε, αυτό που θα ήθελα να μα πει η Κομισιόν όμω, υπάρχει μια απόφαση εδώ, έτσι. Μπορεί κανεί να συμφωνεί, να διαφωνεί, αλλά η απόφαση υπάρχει. Ποιε είναι οι επιπτώσει τη απόφαση, όχι μόνο για τον κλάδο, αλλά και για την έρευνα και την καινοτομία, και για του γεωργού και του καταναλωτέ. Άκουσα κάποιου συνάδελφου να λένε ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ δεν θέλουν την τεχνολογία αυτή. Ε, Βεβαίω αυτό αναφέρεται ω γεγονό. Να προσέχουμε τι λέμε όμω ε, για το τι πιστεύουμε εμεί ότι πιστεύουν οι καταναλωτέ. Ε, πρέπει να ελέγχεται η έρευνα προφανώ. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιε είναι οι επιπτώσει. Όμω εάν επιτραπεί αυτή ε, η μεταλλαξιογέννηση η μία μορφή να επιτρέπεται η άλλη να απαγορεύεται, θέλω να ξέρω γιατί είναι μια επιστημονική συζήτηση δηλαδή που πρέπει να γίνει. Ε, ο καθένας έρχεται με, τις, ε, με το δικό του παρελθόν. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που δεν υπάρχουν γάματα φόμικρον, αλλά τα χρησιμοποιούμε γάματα φόμικρον στις ζωοτροφές. Ε, όπως και περισσότερες χώρες, τα περισσότερα κράτη-μέλη, διότι βασιζόμαστε στην εισαγωγή πρωτεϊνών. Ε, είναι κάτι λοιπόν όπου πρέπει να φανούμε όριμοι στη συζήτηση αυτή. Να καταλάβουμε δηλαδή ποιες είναι οι επιπτώσεις, ο αντίκτυπος της απόφασης και κατά πόσο η νομοθεσία, ε, η υπάρχουσα νομοθεσία είναι κατάλληλη με βάση και την απόφαση του δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, ένα πράγμα είναι σαφές, η απόφαση. Αλλά αυτό που δεν είναι σαφές, εγώ ήμουν σε μια συνεδρίαση της Επιτροπή Γεωργίας για την Αφρική πέρυσι ε, και έθεσα ένα ερώτημα για το γεγονό ότι η Ευρώπη, όταν λέμε ότι η Ευρώπη ταΐζει τον κόσμο, μήπω αυτό είναι κάπως πατερναλιστικό. Και τότε μου είπαν ότι ε, ε, ότι έτσι είναι τα πράγματα, αλλά εγώ μετά κοίταξα στο Google και από ό,τι φαίνεται δεν είναι ακριβώ έτσι. Ε, μιλάμε για χίλιε εκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο ε, στο, στο 2050. Ε, δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη στους ρυθμούς. Θα είναι και μικρότερη. Δηλαδή το γεγονός ε, ότι ε, ταΐζουμε τον κόσμο και ταΐζουμε και ανθρώπους εκτός της Ένωσης, μήπως αυτό είναι πατερναλιστικό, είναι το πιο πατερναλιστικό από όλα, είναι επικίνδυνο που καθιστά τους ανθρώπους εξαρτημένους ενώ δεν πρέπει να είναι εξαρτημένοι. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια είναι η πολιτική της Ένωσης. Θέλουμε να ταΐσουμε τον κόσμο επειδή είμαστε ανώτεροι και μπορούμε, ξέρουμε να το κάνουμε. Ε, αυτό είναι ευρωπαϊκός εθνικισμός. Bardzo Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Όλοι συζήτησαν το λόγο, λοιπόν, να καταφέραν να πάρουν το λόγο. Και άρα μπορούμε να δώσουμε τώρα το λόγο, λοιπόν, στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να απαντήσουν στις παρεμβάσεις και στις ερωτήσεις που έγιναν. Και προφανώ η συζήτηση αυτή συνεχίζεται και σε καμία περίπτωση δεν θα παραμελήσουμε να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Είναι το λόγο λοιπόν. Η Γενική Διευθύνση Υγείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή και που δέλετε το λόγο. Νομίζω ότι αν και δεν ετέθησε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να διευκρινίσω μία πτυχή για μία δήλωση που έγινε από τον βουλευτή του Κρυονιού. Είπατε ότι αν ληφθεί αυτή η απόφαση δεν θα παράγουμε αρκετά τρόφιμα στην Ευρώπη και θα εισάγουμε τα τρόφιμα αυτά. Να διευκρινίσω ότι οι συνέπειες της απόφασης αυτής ισχύουν ανεξάρτητα από το που έχει παραχθεί το τρόφιμο. Είτε πρόκειται για καλλιέργειες εδώ ευρωπαϊκές, είτε πρόκειται για καλλιέργειες που έχουν γίνει αλλού και εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύουν λοιπόν οι ίδιες διατάξεις και ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως προέλευσης των ε, τροφίμων. Και όπως σας είπα αρχικά, Το θέμα διαφοροποίησης ε, των ε, προϊόντων αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί μια πρόκληση θέλουμε να δώσουμε μια απάντηση στο επιστημονικό αυτό ερώτημα και ζητήσαμε από τα εργαστήρια αναφοράς να μας βοηθήσουν από πλευρά των κρατών μελών. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις σε ό,τι αφορά τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων τεχνικών. Και με πάσα ειλικρίνεια θεωρώ ότι είναι υπερβολικό να συζητήσουμε με λεπτομέρεια τις διαφορές των διαφορών τεχνικών. Είναι σαφές ε, το που οδεύει η επιστήμη. Οι νέες μορφές μεταλλαξιογέννησης είναι αυτές που μας ενδιαφέρουν, να ενδιαφέρουν την κοινότητα των ερευνητών, των επιστημόνων, γιατί είναι οι πιο πολλά υποσχόμενες σε ό,τι αφορά το τι αλλαγές μπορούν να γίνουν στην κοινωνική αναπαραγωγή των ε, φυτών σε βάθο χρόνου. Αυτές λοιπόν είναι τεχνολογίες. Το πιο πιστικό ερώτημα είναι, φαντάζομαι, από επιστημονική άποψη για τις τεχνικές αυτές. κυρία Μαγκίνες, ρωτήσατε ποιες είναι πραγματικά οι συνέπειες της δικαστικής απόφασης ε, για την έρευνα και την ανάπτυξη. μπορεί να είδατε τις δηλώσεις ε, των επιστημονικών συμβούλων που εξέτασαν την επιστημονική συνέπεια που θα είχε αυτή η απόφαση και ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Νομίζω ότι η δήλωση της επιστημονικής κοινότητας είναι αρκετά α, αντιπροσωπευτική για το ποιε είναι οι συνέπειε ή ποιε θεωρούν, εν πάση περιπτώσει, οι επιστήμονε ότι θα είναι οι συνέπειε στην έρευνα και την ανάπτυξη και την καινοτομία. Οι συνέπειε τώρα τη απόφαση, αυτό το βλέπουμε και στι διεθνεί συζητήσει. Όχι συνέπεια της απόφασης, αλλά υπάρχουν συνέπειες για το πώς αντιμετωπίζουν οι διεθνείς δικαιοδοσίες αυτές τις νέες τεχνικές μεταλλαξιογέννησης. Εδώ είναι σαφή τα πράγματα. Υπήρχε κάποια σύγκληση σε ό,τι αφορά τους γαματάφ όμικρον, σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες και φαίνεται ότι υπάρχει διαφορετική εκτίμηση στις διάφορες ε, δικαιοδοσίες για το πώς θα ρυθμιστεί αυτό στο μέλλον. Νομίζω ότι δεν είναι ιδιαίτερα προφητικό το να δηλώσουμε ότι θα υπάρξουν συνέπειες ε, σε ό,τι αφορά τη χρήση των τεχνολογιών αυτών στις διάφορες δικαιοδοσίες. Το ανάφερα λοιπόν αυτό και σε ό,τι αφορά τις ε, δικαστικές αυτές αποφάσεις ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση στα προϊόντα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρα ακόμα. Χρειάζεται λοιπόν πιο πολλές πληροφορίες για να δούμε τι θα προκύψει σε ό,τι αφορά και τα επιστημονικά εργαλεία και τα εργαλεία εφαρμογής. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση τώρα να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη για το ποιες θα είναι οι συνέπειες για τους ε, Ευρωπαίους ε, παραγωγούς. Θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο το οποίο έφερα προηγουμένως. σε ό,τι αφορά την ε, βιοτεχνολογία. Ότι θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν αυτή η έρευνα προκειμένου η Ευρώπη να βρει ένα σαφές όραμα για το πού θέλει να οδεύσει στο μέλλον. Εργαζόμαστε στο πλαίσιο το οποίο υφίσταται στην παρούσα φάση, το οποίο ισχύει εδώ για κάποια χρόνια ή κατά πόσον ε, χρειάζεται να εξεταστούν άλλες εναλλακτικέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Ο κύριος Τόρβαλτς θα θέλει να πάρει το λόγο μήπως για να απαντήσει στις παρατηρήσεις που του απευθύνθηκαν για να ικανοποιήσω και το ακροτήριο. Και κυρίως τον κύριο Χόισλινγκ, το φίλο μου. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο σε ό,τι αφορά αυτή την ε, ε, τεχνολογία είναι ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά τεκμήρια που να αποδεικνύουν ότι είναι βλαβερό αυτό ως τεχνολογία. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Ούτε είναι κανείς αντίθετος με αυτά που προασπίζεστε, τη βιώσιμη δηλαδή γεωργία. Και νομίζω ότι εδώ συγκλίνουν οι απόψεις μας σε ό,τι αφορά την βιώσιμη γεωργία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με τεχνολογία ε, αποκοπής τέτοια ε, τμήματων ε, γενετικών. Αυτό που προέκυψε λοιπόν από τη συζήτηση αυτή είναι ότι μπορεί να υπάρχει το ίδιο προϊόν το οποίο να παράγεται από τις παλιές τεχνολογίες γαματάφα όλων μικρών και ένα το ίδιο προϊόν να προκύπτει και με την ε, τεχνολογία αυτή ψαλιδέσματος και το ίδιο προϊόν να προκύψει και με την ε, φυσική εξέλιξη. Δεν είναι όμως σωστός τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης και για το επιχείρημα της βιωσιμότητας εδώ στο, στη συζήτηση αυτή εφόσον το δικαστήριο έχει λάβει απόφαση. Εμείς είμαστε σε θέση να την επικρίνουμε την απόφαση αυτή. Αυτή είναι η δημοκρατία. Τα σχόλια του ότι «Α, εφόσον ελήφθησε η δικαστική απόφαση δεν έχουμε δικαίωμα να το συζητάμε καν», θεωρώ ότι αντιβαίνουν στην αρχή της δημοκρατίας. Θα πρέπει να μην προσπαθείτε να περιορίσετε το δικαίωμά μου να συζητώ μια απόφαση του δικαστηρίου. Υπάρχει μια αφαία ε, περιοχή, μια γκρίζα τέτοια με κρίσεως τομέας, όπου τίθεται και επιστημονικό ζήτημα. Σας παρακαλώ λοιπόν να επιδεικνύετε τον απαραίτητο σεβασμό. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι αυτή ήταν ε, μια πολύ καλή ολοκλήρωση των συζητήσεων που ε, έλαβαν χώρα. Εδώ ε, θέλουμε να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων και αυτό δεν είναι ενδιαφέρον εάν όλοι έχουν την ίδια άποψη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ξέχασα τον κύριο Άγνιο που είχε ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, με ανέφερε με το όνομά μου η ε, εκπρόσωπος της Κομισιόν. Εάν δούμε τι έχει συμβεί με τα ε, μεταλλαγμένα, 30.000 τόνους εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο ε, και βεβαίως εάν ταξινομούμε τις, τις με τον ίδιο τρόπο αυτές, με τις οδιές με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ταξινομούμε τις κανονικές σοδιές, τότε θα έχουμε έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και πρέπει να σας πω ότι καμιά φορά μέσα από μια διαδικασία που στην αρχή φαίνεται αμφιλεγόμενη μπορεί να προκύψουν ποικιλίε τις οποίες χρησιμοποιούμε όλοι ε, και ε, η παραγωγή με μεγάλη ευχαρίστηση τις χρησιμοποιούν. Ευχαριστώ πολύ. Ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Όχι. Επομένω μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Όπως ε, είπα και προηγουμένω οπωσδήποτε δεν είναι η τελευταία συνάντηση και η τελευταία συζήτηση. Άλλωστε ούτε και η κοινωνία ε, δια των εκπροσώπων της δεν είναι σύμφωνη, δεν έχει την ίδια άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, στις 14 Ιανουαρίου θα λάβει χώρα η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας και αυτό θα γίνει στο Στρασβούργο. Αυτά για σήμερα και ολοκληρώθηκε η συνεδρίασή μας. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Α, συγγνώμη, η κυρία Αγγιλέρα θέλει το λόγο. Muy brevemente, señor presidente. Ε, ναι, Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Ε, επειδή είναι η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής το 2019, ήθελα να αναφέρω κάτι για τη συμφωνία για τα σπυριδοειδή με την Νότια Αφρική. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Με αυτήν την ε, επέκταση στις έξι εβδομάδες αυτό θα πέσει πάνω στην εκστρατεία, πάνω στη σοδεία μάλλον, ε, πρέπει να γίνει μια συζήτηση, το έχω προτείνει και στους συντονιστές της Επιτροπής μας, να γίνει μια συζήτηση λοιπόν για την εφαρμογή, ειδικά της, εφαρμογή, της ε, συμφωνίας με την Νότια Αφρική και την ζημιά που προκαλείται για τους ε, καλλιεργητές περιδοειδών της Ευρώπης κυρίως ιδιαίτερα της χώρας μου της Ισπανίας. Ήθελα να το πω στο τέλος για να συζητηθεί στη συνδέα των συντονιστών. Ευχαριστώ. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος, θα ζητήσουμε από την ε, Γραμματεία να το εντάξει ε, κάπου. Θα το συζητήσουμε στους συντονιστές και μετά ε, στην κανονική συνεδρίαση της ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς. Καλό βράδυ. Πολύ ωραία ξεκίνησε η νέα χρονιά με εντατικές και ωραίες εργασίες. Ευχαριστώ.